Um, λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Θα συζητήσουμε ποινικέ κυρώσει για τι πράξει προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικέ πληροφορίε και τι πράξει χειραγώγηση αγορά. Η κυρία Βοσκούρη είναι η λέει ότι οδηγεί η κατάχρηση της αγοράς του 2003 παρά το ότι σιγάγει ένα πλήρες πλαίσιο για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο που προανέφερα δεν πέτυχε το στόχο να αυξήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και την ακεραιότητα της αγοράς. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέο νομικό πλαίσιο που συμπεριλαμβάνει μια πρόταση οδηγίας για ποινικέ κυρώσεις για το όλο φαινόμενο και προτείνεται και κανονισμό για το ίδιο φαινόμενο. Η Επιτροπή Ελευθεριών μοιράζεται τι αρμοδιότητες στην Επιτροπή την Οικονομική, σύμφωνα με το άρθρο 50, αλλά από ό,τι φαίνεται το θέμα του επιμερισμού των αρμοδιοτήτων δεν έχει οριστικά επιληθεί από τη διάσκεψη των Προέδρων. Γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις αλλά εν τω μεταξύ ε, μας εμποδίζει, δεν μας εμποδίζει να συζητήσουμε πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις 21 Απριλίου παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ακούσουμε την κυρία Μποσκούρ την εισηγήτρια, τι έχει να μας πει. Και να σας πω ότι η προθεσμία για την υποβολή ε, τροπολογιών είναι το μεσημέρι της 5ης ε, Ιουνίου. Κυρία Μποσκούρ, ευχαριστώ πάρα πολύ όσον αφορά το θέμα αυτό, την πρόταση αυτή. Λοιπόν, οι κυρώσεις εξετάζονται για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Η οδηγία για την τη αγοράς του 2003 δεν έχει πετύχει το στόχο, την αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και την ακεραιότητα της αγοράς, όπως είπε και η Πρόεδρος. Δεν έχει λοιπόν επίδραση και δεν είναι αρκετά αποτρεπτική, άρα Αποτελεσματική είναι η επιβολή της οδηγίας. Πέραν αυτού, ο ορισμός όσον αφορά την κατοχή πιστωτικών πληροφοριών και τις πράξεις της αγοράς και πώς μπορούν αυτές να θεωρηθούν ποινικά δικήματα, η ερμηνεία ποικίλει από χώρα σε χώρα. Αυτή η απόκληση υπονομεύει την εσωτερική αγορά και αφήνει και κάποιο πεδίο δράσης για εκείνους που θέλουν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Οι ποινικέ κυρώσεις για τις σοβαρότερες, τις σοβαρότερα αδικήματα είναι πολύ, ε, κάτι πολύ χρήσιμο ούτω ώστε να εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι πολιτικές ε, της Ένωσης όσον αφορά την ε, τη χειραγώγηση αγοράς. Άρθρο 83.2 είναι η βάση που χρησιμοποιείται και πρέπει να θεωρηθεί σαν πακέτο που συμπεριλαμβάνει και την πρόταση κανονισμού όσον αφορά τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και τη χειραγώγηση της αγοράς. Εκεί δεν έχουμε κοινή αρμοδιότητα και η Οικονομική Επιτροπή ασχολείται με το θέμα. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται συνέπεια μεταξύ των δύο νομικών μέσων. Τι συνεπάγεται αυτό, ότι οι ορισμοί των διοικητικών και ποινικών αδικημάτων θα πρέπει να είναι κάτι συνεπές. Ταυτόχρονα θα πρέπει να σεβόμαστε και την αρχή της ασφάλειας δικαίου περιγράφοντας τα στοιχεία που αποτελούν το ποινικό αδίκημα όσο ακριβέστερα γίνεται, τόσο ώστε τα άτομα να μπορούν να καταλάβουν επακριβώς ποιες δράσεις καταστούν αυτούς ποινικώ ε, διώξιμους και υπεύθυνου. Γι' αυτό για τα άρθρα και 4 έχω αποβάλει τροπολογίες ε, και για την τα αποτρεπτικά μέτρα του ποινικού δικαίου δεν θα πρέπει να ειδωθούν από τα ΜΜΕ να, αποτελείται, να είναι αποτρεπτικό παράγον η προβολή στα ΜΜΕ, αλλά τα ίδια τα μέτρα είναι αποτρεπτικά και θα πρέπει να υπάρχουν και διάφορα δικαιώματα που έχουν οι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στι διάφορε διαδικασίε, στι δίκε. Αυτό το αναφέρω στι ιδεολογικέ σκέψει. Μετά έχουμε την αρχή της, του Nebis ε, in idem, δηλαδή ε, να μην δικάζεται δύο φορές κάποιος, δύο φορές το ίδιο ε, υπάρχουν και ανησυχίες για το ισχύον ε, καθεστώς που είναι τερογενές, θα πρέπει μέχρι τις κυρώσεις να εναρμονιστούν. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο ενδεδειγμένο σαν μέτρο. Θα σταματήσω εδώ και θέλω να ακούσω τι θα μας πούν το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Ρατκόφσκι για το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά το θέμα αυτό, σας λέω ότι εκφράζω την άποψη του κυρίου Σόνικ, ο οποίος δυστυχώς δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στη συνεδρίασή μας. Θέλω να πω λοιπόν το εξή ότι η οδηγία θέσπισε ένα πλαίσιο πλήρες όσον αφορά την κατοχή εμπιστευτικών πληροφοριών και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, δεν αυξάνει όμως την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην αγορά. Νομίζω ότι βασικός λόγος γι' αυτό ήταν ότι οι κυρώσεις που προβλεπόταν δεν ήταν αρκετά αποτρεπτικές. Εν γέννη, διάφορα κάτι μέλη καθορίζουν διαφορετικά Ποιε τέτοιε πράξει όπω ε, χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών θεωρούνται ποινικά κολάσιμε. Η χειραγώγηση τη αγορά μπορεί να έχει διεθνή εμβέλεια και μπορεί να είναι επιβλαβέστατη και να εμποδίζει τη λειτουργία εσωτερική αγορά. Υπάρχουν διαφορέ στα διάφορα κράτη-μέλη όσον αφορά τι ποινικέ κυρώσει και αυτό υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά. Και αυτοί που διαπράττουν αυτέ τι πράξει ε, δεν μπορούν να δικαστούν κανονικά και μπορούν να βρουν τα συστήματα εκείνα τα οποία είναι τα πιο ελαστικά και τα πιο επίκη. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το καταργήσουμε και να θεσπίσουμε πραγματικά αποτρεπτικές κυρώσεις. Το παρόν πλαίσιο δεν προβλέπει σωστές κυρώσεις, άρα συνεπάγεται λογικός ότι θα πρέπει να προβούμε σε ελάχιστη εναρμόνεση των κυρώσεων και πρέπει να θεσπίσουμε ελάχιστου κανόνε όσον αφορά τη χειραγώγηση τη αγορά και τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών. Αυτού του είδου η δραστηριότητα θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση τη εμπιστοσύνη των επενδυτών και θα πρέπει να εισαγάγει και κάποια σταθερότητα στι χρηματοπιστωτικέ αγορέ. Όσον αφορά τι τροπολογίε, νομίζω ότι θα πρέπει να καθορίσουμε πόσα έτη φυλάκιση θα είναι κύρωση για κάποιον που διαπράττει αυτού του είδους το έγκλημα και περιορισμός των της σε δύο ή πέντε χρόνια δεν είναι καλή ιδέα. Πιστεύουμε ότι οι ποινικέ κυρώσεις θα πρέπει να θεσπίζονται χωρίς να τίθεται ανώτατο όριο ε, για συγκεκριμένο έγκλημα. Διαφορετικά δικήματα ε, κολλάζονται με διαφορετικές ποινές και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν και τα κράτη-μέλη εκείνα που δεν έχουν θεσπίσει μέχρι τώρα ποινές θα μπορέσουν να το κάνουν παίρνοντας σωστές αποφάσεις, ποινικοποιώντα αυτού του είδους τις πρακτικές στο μέλλον. Νομίζω το άρθρο 3 θα πρέπει και αυτό να ολοκληρωθεί. Αναφέρεται στη χρήση εσωτερικών εμπιστευτικών πληροφοριών. Θα προσθέσουμε, θα προσθέσουμε και άλλο στοιχείο. Να ποινικοποιούμε τις πράξεις εκείνου που προσπαθεί μέσω άλλου ανθρώπου να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα μέσα της αγοράς εκμεταλλευόμενος εμπιστευτικές πληροφορίες. Insider dealing. Αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ε, και ως ε, ότι γίνεται συνεργός αυτό στη διάπραξη της πράξης. Αλλιώς, εάν βάλουμε ανώτατο όριο στο ποινικό μας σύστημα και άλλο ένα όριο, αυτό θα αποδυναμώσει την όλη προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Οπότε να ακούσουμε την Κομισιόν, την κυρία Ζουλ Σχέντερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια κυρία Μποσκούρτ για την έκθεσή της. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή σας δηλαδή και η Επιτροπή συμμερίζομαστε έναν κοινό στόχο, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο για να αποφύγουμε τις παράνομες αυτές πρακτικές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ώστε να εξασφαλιστεί η ακαιρεότητα των αγορών και η ασφάλεια των επενδυτών. Άρα είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. Θέλω να σα ευχαριστήσω και για τι επικοδομητικέ σα τροπολογίε. Κάποιε παρατηρήσει από πλευρά μα θα ήταν οι εξή. Πρώτα απ' όλα, Υπάρχει πράγματι το ζήτημα αυτό της συνεκτικότητας που ανέφερε η κυρία Μποσκούρτ για την ε, χειραγώγηση της αγοράς, τον κανονισμό και την οδηγία για ποινικέ κυρώσεις σε περίπτωση χειραγώγησης της αγοράς. Θα πρέπει να δούμε τους ορισμούς ε, και το πεδίο, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια. Θα επανεξετάσουμε τα σχετικά και μελετάμε με πολύ προσοχή τις τροπολογίες σας. Για να δούμε ακριβώς τι γίνεται και με τα δικαιώματα και στις δύο περιπτώσεις. Για τις κυρώσεις, να πω κάποια πράγματα, η πρόταση της Κομισιόν δεν προβλέπει μια κατώτατη ή ανώτατη κύρωση και αυτό για αρκετούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νομικό μέσο βάσει του άρθρου 83 παράγραφος 2. Αυτό αποτελεί νεοτερισμό στο πεδίο του ποινικού δικαίου. Άρα αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με μια προσεκτική προσέγγιση. Αυτό είναι ένα πρώτο επιχείρημα και ένα δεύτερο, ένα σημαντικότερο επιχείρημα είναι ότι δεν έχουμε ακόμη μια πλήρη εικόνα για τις πρακτικές των κρατών μελών, δηλαδή σε ό,τι αφορά το εθνικό ποινικό δίκαιο που ισχύει αυτή τη στιγμή, Άρα δεν μπορούμε και να καθορίσουμε κατόφλια, είτε για την ανώτατη για την κατώτατη κύρωση, σε περίπτωση χειραγωγής αγοράς. Πάντως, πιστεύουμε και εμείς ότι εν τέλει καλό θα ήταν να υπάρχει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο και για τις κυρώσεις, έξω και στην πρότασή μας λέμε ότι θα πρέπει να γίνεται μια έκθεση για την εφαρμογή της ε, οδηγίας αυτό η έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί σχετικά σύντομα, ώστε να δούμε πώ εφαρμόζεται το μέσο αυτό από τα κράτη-μέλη και να δούμε τι θα κάνουμε και με τι κυρώσει. Τελευταίο σημείο, το νέμπι νίντεμ, το διπλό αξιόπινο δηλαδή, που λέει και η κυρία Μποσκούρτ. Είναι προφανές ότι θα πρέπει η πρόταση αυτή να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αρχή του νέμπι νίντεμ, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην συγχαίουμε το διπλάξιο πνεύμα και τη σχέση μεταξύ ποινικών και διοικητικών κυρώσεων. Γιατί κάποιες φορές με τις διοικητικές κυρώσεις δεν ε, ε, ενεργοποιείται η αρχή του νέμπις in idem. Πρέπει να υπάρχει και ένα ποινικό στοιχείο. Τα κράτη-μέλη βέβαια είναι αυτά τα οποία θα έχουν την ευθύνη γιατί πρέπει να δούμε πώς εφαρμόζουν τις ποινικές κυρώσεις και πόσες διοικητικές κυρώσεις και μετά θα δούμε στο τέλος πώς μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το θέμα. Πρόεδρος. Έφτασε και ο κ. Διόν και προφανώς θέλει και αυτό το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και θα πρέπει να πω ότι δεν θα κάνω σχόλια επί των λεπτομεριών, επί των επιμερών στοιχείων. Να πω όμως ότι στην προηγούμενη Ολομέλεια ε, ψηφίστηκε η έκθεσή μου για το ποινικό δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα από τα θέματα που τέθηκε πέρα από την συνοχή και τη συνεκτικότητα είναι ότι θα πρέπει να πιστούμε ότι ο μοναδικός τρόπος να προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τα μέσα ποινικού δικαίου είναι μια ποινική προσέγγιση, να δούμε τεκμήρια της ανάγκης αυτή και επίσης ε, την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή προσέγγιση. Να πω ότι γενικά δεν είχα προβλήματα με την ε, πρόταση, αλλά θα πρέπει να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά και γι' αυτό ρωτάω και την εισηγήτρια και την Επιτροπή πώς θα αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό, πού μπορώ να διαβάσω τα κριτήρια τα οποία έχει εγκρίνει προσφάτως το Κοινοβούλιο, να δω ότι, έχουν, ε, ότι πληρούνται στην προκειμένη περίπτωση. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, και αν δεν θέλει να σχολιάσει καμία, κανένας άλλος ε, ε, συνάδελφος, να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για να κάνει καταληκτικά σχόλια. Ναι, σας ευχαριστώ. Άκουσα. Δεν ξέρω το συμβούλιο, μήπως θα πάρει το λόγο πρώτα. Το Συμβούλιο δεν αποφάθηκε. Όχι, με ενημέρωσαν, λέει ο Πρόεδρο, ότι το Συμβούλιο δεν ε, επιθυμεί να πάρει το λόγο. Α, μάλιστα, δεν το κατάλαβα, λέει η συγγήτρια. Σα ευχαριστώ, όπω και να έχει, για, την... Ε, για το feedback. Να μιλήσω Ολλανδικά. Δύο ερωτήσει είχα να κάνω μετά από τις παρεμβάσεις ε, και προς τον συνάδελφο του ΕΛΚ να πω ότι θεωρώ ότι κινούμαστε στις ίδιες γραμμές λίγο πολύ. Ίσως να υπάρχει κάποια διάσταση απόψε για την επιβολή κυρώσεων. Το θέμα για όλη αυτή την οδηγία, τι προσπαθούμε να βελτιώσουμε. Αυτό που έχουμε, καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι δεν λειτουργεί όταν μιλάμε για την χειραγώγηση αγοράς, αυτό είναι κάτι το οποίο κινείται διασυνοριακά, γιατί αυτοί που κάνουν τη χειραγώγηση της αγοράς ε, ξέρουν να εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες του συστήματος και να πάνε στη χώρα που δεν πρόκειται να τους πιάσουν. Άρα, τη στιγμή που θα αφήσουμε τα κράτη μέλη να καθορίσουν ποια θα είναι τα ελάχιστα πρότυπα, το πρόβλημα θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Γιατί πολύ απλά θα πηγαίνουν οι ύποπτοι στις χώρες αυτές με τα ε, χαμηλότερα πρότυπα. Δεν ξέρω κατά πόσο να έχει νόημα να αφήσουμε έτσι την διάταξη αυτή. Προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ρωτήσω το εξή. Για το διπλό αξιόπινο. Σωστά καταλαβαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι είναι προβληματικό κάποιος ο οποίος έχει ε, κατηγορηθεί και καταδικαστεί για πράξεις χειραγώγησης της αγοράς θα πρέπει να λάβει διοικητικές κυρώσεις αλλά και ποινικές κυρώσεις. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι προτείνεται. Καταλαβαίνω ότι στην πράξη κυρίως ποινικές είναι οι κυρώσεις που επιβάλλονται. Αλλά σας παρακαλώ, γιατί ευκρινίστε τι εννοείτε. Αυτά ήθελα να πω λοιπόν μετά τις παρεμβάσεις που ακούσαμε. Η Πρόεδρος, μάλιστα. Επειδή δεν έχουμε τόση χρονική πίεση όσο συνήθως, να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει εν συντομία. Γιατί πάντα λέω ότι σκοπός μας δεν είναι να ε, γεμίσουμε το χρόνο μας μέχρι τις 6.30. Ευχαριστώ πολύ για την τροπολογία 8 και τη σχέση μεταξύ διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. Η διατύπωση, όπως προτείνεται από την κυρία Μποσκούρτ, θεωρούμε ότι είναι κάπως αυστηρή, γιατί όταν έχουν επιβληθεί διοικητικέ ε, κυρώσει αποκλείεται η πιθανότητα επιβολή ποινικών κυρώσεων. Οι διοικητικέ ε, και ποινικέ κυρώσει εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο στα κράτη-μέλη. Κάποια κράτη-μέλη μπορούν να τις εφαρμόσουν και τις δύο κυρώσει. Καταλαβαίνουμε μεν ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο υποβλήθηκε η τροπολογία και φυσικά είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε για την εκ νέου διατύπωση της τροπολογίας προκειμένου να επαφείεται στο σύστημα του κράτους μέλους το πώς θα δρά. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον δυνατότητα εφαρμογής ποινικών κυρώσεων, ακόμα και αν έχουν ήδη επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο και τελευταίο σημείο για την ημερήσια διάταξη για σήμερα. Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν για την περίοδο 1 1η Νοεμβρίου 2011 μέχρι 30 Απριλίου 2012. Πρόκειται για την πρώτη σε έκθεση, αλλά νομίζω ότι είναι εξαμηνία η έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν. Η Επιτροπή δεν έχει καταφτάσει ακόμη, λέει η Πρόεδρος. Λίγα λεπτά διάλειμμα τότε, μέχρι ότου καταφτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Um, colleagues, I think that uh, <laughs> the Commission is here now. Συνάδελφοι, νομίζω ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε και δύο ακριβώς βουλευτές μαζί μας. Οι τελευταίοι του Μαϊκανών. I'm looking at the staff. Coelho's coming? Okay, I think it's worthwhile to wait for Mr. Coelho. Να περιμένουμε τον κύριο Coelho. Λίγα λεπτά ακόμα υπομονή σας ζητώ. Γιατί είναι κρίμα να είμαστε τόσο λίγοι και να μην χρειάζεται να πάρουμε οποιοδήποτε απόφαση. Φανταστείτε τι θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε. Okay, Συνάδελφοι, τώρα που μαζευτήκαμε όλοι, σας ευχαριστώ και για την υπομονή σας. Το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διαταξή τη σημερινή, να δώσω το λόγο στην κυρία Μελίντα Πλέικ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. μεγάλη μου χαρά Ήρθα στο Κοινοβούλιο σήμερα για να σας δώσω μια συντομή επισκόπηση για μια έκθεση την οποία ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Μαΐου στην εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν 1 ε, Νοεμβρίου του 2011, 30 Απριλίου 2012. Στα αγγλικά έγινε η έγκριση. Ελπίζω να έχετε όμως και τις υπόλοιπες γλώσσες για τους βουλευτές να εξηγήσω και ποιο είναι το υπόβαθρο της έκθεσης, να πω δύο λόγια για τα στοιχεία που περιλαμβάνει και να πω και δύο λόγια για τα επόμενα βήματα και η Προεδρία και αυτή θα πει δύο λόγια για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει το θέμα αυτό στην συνάντηση του Συμβουλίου την επόμενη Πέμπτη. Γιατί έγινε λοιπόν αυτή η εκθέση. Όπως ξέρετε είμαστε στο 27ο έτος του Σέγγεν. Το σύστημα λειτουργεί καλά, αλλά υπόκειται πιέσει. Ε, και όπως όλα τα συστήματα, πρέπει να το παρακολουθούμε για να βεβαιωνόμαστε ότι λειτουργεί σωστά. Στην ανακοίνωσή μας ε, το, το προηγούμενο Σεπτέμβριο για την ενίσχυση του Σέγγεν, θέλαμε να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα. Δύο εξ αυτών είναι νομοθετικά. Ε, μηχανισμός ε, αξιολόγησης και άλλα, ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε και από την Επιτροπή σας, η ανακοίνωσή σας, αυτή πρότεινε να ε, γίνει και ένα health check κάθε έξι μήνες να γίνεται για το χώρο Σέγγεν και σκοπός της πρότασης αυτής είναι να δώσουμε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τη δυνατότητα να εξετάσουν τακτικά τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν. Και τώρα θα ήθελα να πω δύο λόγια για την ίδια την έκθεση. Καταρχάς, σκεφτήκαμε πολύ το πεδίο εφαρμογής. Και σκεφτήκαμε και άλλες ε, εκθέσεις που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση. Για παράδειγμα, την ετήσια έκθεση για την ε, μετανάστευση και το άσυλο που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα θεωρήσαμε ότι αυτές ήταν σχετικά τα θέματα αυτά. Στην ίδια την έκθεση εστιαζόμαστε σε μια σειρά θεμάτων. Καταρχάς την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα. Και εκεί, όπως τονίζουμε, η πίεση στα εξωτερικά σύνορα ε, εστιάζεται σε κάποια ε, σημεία στην Ανατολική Μεσόγειο, κυρίως και Νότια Μεσόγειο. Και συνεχίζουμε να αξιολογούμε τα μέσα με τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τα κράτη-μέλη στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, αλλά ασφαλώς παραμένουμε ανοιχτοί στις ε, παρατηρήσεις ε, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το κατά πόσον ε, υπάρχει ισορροπία στα μέσα αυτά και φυσικά περιμένουμε και σχόλια. Ο δεύτερος τομέας είναι οι ροές μετανάστευσης, οι ροές κίνησης στο χώρο Σέγγεν και αυτό είναι πάρα πολύ επίκαιρο θέμα. Είδαμε τα αποτελέσματα επιχειρήσεων, δράσεων που διοργανώθηκαν από διάφορες προεδρίες και προσφάτως από την Δανική Προεδρία και από την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία για την αξιολόγηση της κατάστασης. Όπως εξηγούμε στην έκθεση, δυστυχώς δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη στις δράσεις αυτές και θεωρούμε ότι αν το έπραταν αυτό, τα στοιχεία θα ήταν πιο αξιόπιστα, θα είχαμε πιο τεκμηριωμένα στοιχεία για τις δευτερεύουσες ε, ε, μεταναστευτικές ροές στο χώρο Σέγγεν και νομίζω ότι με τέτοιες πληροφορίες θα μπορέσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να λάβει ενημερωμένη απόφαση, ενημερωμένες αποφάσεις ε, για τα προβλήματα που εντοπίζονται. Ένας τρίτος τομέας, τον οποίο εξετάζουμε στην έκθεση, είναι η εφαρμογή του κεκτημένου. Και στο σημείο αυτό συνοψίζουμε κάποια μέτρα για την ε, παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας των σχετικών μέτρων στα κράτη-μέλη και φυσικά και ενδεχόμενες ε, ενστάσεις που λαμβάνουμε καταγγελίες από τους πολίτες. Και πολλές είναι οι ανησυχίε που εκφράζονται από πολίτες, από οικονομικούς φορείς σχετικά με μέτρα τα οποία λαμβάνουν τα κράτη-μέλη, τα οποία ενδεχομένως να θεωρούνται έλεγχος εσωτερικών συνόρων. Επίσης τονίζουμε τους τομείς στους οποίους ένα κρατός μέλος χρησιμοποιεί τα δικαιώματα τους ε, υπό το χώρο Σέγγεν για να επανεισάγει εν μέρη συνοριακούς ελέγχους, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία πρόσφατα σε ό,τι αφορά την Κεντρική Τράπεζα και ξέρουμε ότι σε σχέση με το ποδοσφαιρικό στις ποδοσφαιρικές εκδηλώσεις ε, ότι οργανώνονται, μάλλον επανεισάγονται σχετικές, ε, σχετικοί έλεγχοι στην Πολωνία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σύστημα πληροφόρησης Schengen, θεωρούμε ότι το σύστημα αυτό ε, χρήση κάποιων βελτιώσεων. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ χρήσιμο και πολύτιμο εργαλείο για τα κράτη-μέλη και ε, θεωρούμε από τις συζητήσεις μας με τα κράτη-μέλη ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά το σύστημα προκειμένου να μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι κάθε κράτος μέλος χορηγεί τις πληροφορίες και το σύστημα Siren μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω προκειμένου να μην υπάρχει ε, καθυστέρηση όταν ένας νοριοφύλακας επιθυμεί να μάθει πιο πολλά για πληροφορίες που χορηγήθηκαν από άλλο κράτος ε, μέλος. Ε, το σύστημα πληροφόρησης θεωρήσεων που ξεκίνησε πρόσφατα και να σας πω ότι από τότε που συγγνώμη, εισήχθη το σύστημα VIS ε, έχει χρησιμοποιηθεί πολύ από τα κρατη και τα επόμενα χρόνια θα εισαχθεί και σε, άλλους, ε, σε άλλα μέρη. Τέλος, το θέμα της πολιτικής θεωρήσεων και της επανεισδοχής. Ξέρουμε ότι το θέμα των θεωρήσεων επηρεάζει και τις αιτήσει ασύλου στη Σουηδία, για παράδειγμα στο Βέλγιο, σε ό,τι αφορά τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και θέλουμε να ακούσουμε και τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ξέρω και ότι το Συμβούλιο θα το συζητήσει το θέμα αυτό την επόμενη εβδομάδα. Επίσης να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε καθεδρίες γραμμές για τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν. Ανακοινώσαμε ότι αν χρειαστεί θα καταρτήσουμε τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές για θέματα εθνικών αρμοδιοτήτων που άπτονται όμως του χώρου Σέγγεν. Οι κατευθυντήριες γραμμές που καταρτήσαμε μετά από διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες περιλαμβάνουν ε, αστυνομικά ζητήματα, στα ιστορικά σύνορα, έχουν να κάνουν μεταξυβετικά έγγραφα και το καθεξής. Θεωρούμε ότι είναι χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες για κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την άσκηση των εθνικών τους αρμοδιοτήτων στο χώρο Σέγγεν. Καλωσορίζουμε ορίζουμε τις απόψεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την επόμενη εβδομάδα το Συμβούλιο θα συζητήσει τα θέματα αυτά στις 7 Ιουνίου και Χαίρομαι που η Προεδρία θα μας πει δύο λόγια για την επερχόμενη αυτή συζήτηση. Η επόμενη έκθεση το Νοέμβριο για την εξαμηνία περίοδο. Ελπίζουμε και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο με τον τρόπο αυτό να λαμβάνουν τακτικά μία επισκόπηση για το πώς λειτουργεί ο χώρος Σέγγεν μετά από 27 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ Στρέφομαι προς την Προεδρία του Συμβουλίου. Ο κύριος Ανκαστιένε, εκπρόσωπος της Δανικής Προεδρίας, συγγνώμη αν δεν πρόφερα σωστά το όνομά σας, πολύ σωστά το... Μία από τις καλύτερες ε, φορές που είπαν το όνομά μου. Λυπάμαι που έχω τόσο περίπλοκο όνομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχτήκατε εδώ ε, και ευχαριστώ για την ωραία παρουσίαση της νέας έκθεσης. Πράγματι είναι πολύ σύντομη, περιεκτική. Περιγράφει πολύ σωστά την κατάσταση κατά την άποψή μας και αναφέρει και ενδεχόμενε πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την συνεργασία στο Σέγγεν. Είναι προφανές ότι ενισχυμένη και βελτιωμένη προσέγγιση στον αφορά το Σέγγεν, ένα βελτιωμένο σύστημα, θα εξασφαλίζει ακόμα καλύτερο έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και αυτό συνδέεται και πολύ με το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης. Αν δεν υπάρχουν ασφαλή εξωτερικά σύνορα, δεν θα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα για την ελεύθερη μετακίνηση εντός του χώρου Σέγγεν. Τα συμπεράσματα της 8ης Μαρτίου του Συμβουλίου έλεγε ότι, έλεγαν ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να είναι η βάση μαζί με συστάσεις για στρατηγικές συζητήσεις στη Μικτή Επιτροπή σε υπουργικό επίπεδο τον Ιούνιο. Σύμφωνα λοιπόν με τα συμπεράσματα προγραμματίσαμε συζήτηση που θα λάβει η χώρα στα περιθώρια του Συμβουλίου που θα γίνει στις 7 και 8 του Ιουνίου. Συμβουλίου Δικαιοσύνη. Η έκθεση είναι πολύ καλό υπόβαθρο για τη συζήτηση και η σημερινή συνάντηση και αντιδράσει των μελών της Επιτροπής σίγουρα επίσης θα τροφοδοτήσουν και θα βελτιώσουν τις συζητήσεις στο Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Επιλέγουμε σε αυτή τη φάση τα θέματα προς συζήτηση και ένα θέμα το οποίο θεωρούμε προφανές είναι μια αναθεώρηση που συνέστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιους θερμούς τομείς, αν δίνουμε επαρκή υποστήριξη, αν εστιαζόμαστε στα προβληματικά σημεία, μήπως πρέπει να υποστηρίξουμε κάποιους τομείς ε, που ήδη θεωρούνται προβληματικοί ή να βρούμε νέα σημεία προβληματικά. Αυτά είναι ένα από τα θέματα προς συζήτηση στο συζητήση Συμβουλίου. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Μέχρι τώρα πρέπει να πούμε ότι όλοι οι παρόντες θέλουν να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Κοέλιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα, θα ήθελα να πω λοιπόν ότι ξεκινώ ευχαριστώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υποβάλλει αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση αυτό το έγγραφο για τη διακυβέρνηση του Σέγγεν, του φόρου Σέγγεν ε, θα συζητείτε τακτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μάλλον θα υποβάλλονται εκθέσει τακτικά στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, ζώνη Σέγγεν. Έγινε αυτό πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε που μα υπέβαλε την έκθεση. Είναι σαφή, σύντομη, περιεκτική και τα βασικά σημεία που αφορούν το θέμα Σέγγεν εμπεριέχονται και είναι καλά και τα παρατήματα. Θα πρέπει να καταλάβετε, Πρόεδρε, όμως ότι θα πρέπει να τονίσω ότι είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι μέσω της πρωτοβουλίας αυτής δείχνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θεωρεί ότι είναι κρίσιμος και σημαντικός εταίρος το Κοινοβούλιο για τη συζητήση για το Σέγγεν. Είναι μια στάση σεβασμού έναντι του Κοινοβουλίου θα έλεγα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέρη εποφελώς, όλα τα θεσμικά όργανα. Μετά θέλω να πω ότι φαίνεται ότι το πακέτο Σέγγεν είναι κάτι σημαντικό και προβλέπει και την υποχρέωση αυτής της ενημέρωσης. Το πακέτο Σέγγεν διακυβέρνηση του Σέγγεν αποτέλεσε αντικείμενο πολλών πρωτοβουλειών που συζητούνται ακόμα. Μόνο όμως αυτή η δέσμευση τελικά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται να μεταφράζει τις προτάσεις που είχαν αρχικά εισαχθεί στο πακέτο σε πράξη. Τρίτον, θα ήθελα να επαναλάβω ότι για όλους εκείνους που δίνουν μία αξία, μία σημασία στο θέμα, η επέκταση του Σέγγεν και η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών είναι κάτι που αφορά τα συμφέροντα τα κοινοτικά και συμφέρουν την κοινότητα. Γνωρίζουμε ότι σε αυτό το τομέα υπάρχει ειδική ευθύνη των κρατών μελών που έχουν αρμοδιότητα παραπόνα να εγγυώνται ε, την προστασία από πλευράς τους του δικού τους κομματιού των εξωτερικών συνόρων. Αλλά είναι σαφές ότι το Σέγγεν δεν είναι αρμοδιότητα. Είναι μια ευθύνη. Πρέπει να είναι μια κοινοτική ευρωπαϊκή ευθύνη το Σέγγεν. Οπότε θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μία ένταση μεταξύ εκείνων που πριν από τη Λισαβόνα θεωρούσαν ότι ήταν κάτι διακυβερνητικό και από την άλλη υπάρχουν εκείνοι όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τώρα θεωρούν ότι είναι σαφώς μια ευρωπαϊκή διάσταση που θα πρέπει να γίνει σεβαστή. Αυτή η ανακοίνωση που παραλάβαμε, σύμφωνα με την οποία η Προεδρία παρουσίασε στο Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό μια πρόταση τροποποίησης της νομικής βάσης ε, του συστήματος αξιολόγησης Σέγγεν, ούτω ώστε να, να αφαιρεθεί η συναπόβαση από το Κοινοβούλιο, που έτσι δεν θα μπορούσε να ε, συμμετέχει σε μια σημαντική ε, διάσταση την αξιολόγηση του Σέγγεν. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία που αντιστοιχεί στροφής προς διακυβερνητική οπτική γωνία που απομακρύνεται από την κοινοτική προσέγγιση. Λοιπόν, Πρόεδρε, αναλύοντας την έκθεση, χαιρετίζω το περιεχόμενο, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρωτοβουλία αυτή, όμως ε, καταγγέλλω αυτές τις τελευταίες εξελίξεις στο Συμβούλιο. Λυπάμαι γι' αυτός. Και θα ζητούσα μάλιστα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει Όσον αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση του Σέγγεν, τώρα, αν είναι εξίσου απεσιόδοξη όπως εγώ και όπως πιστεύω όλοι μας εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Έντσου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την πρώτη έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν. ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας ε, παρουσίασε αυτή την έκθεση με απόγευμα. Η έκθεση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο να συζητούμε σοβαρά το θέμα το οποίο είναι τόσο σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζω ότι τα κράτη-μέλη και εκείνα θα, λάβουν, θα χρησιμοποιήσουν τον χρόνο τον αναγκαίο για να αναλύσουν την έκθεση και να συναγάγουν τα συμπεράσματά τους και ελπίζω ότι θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα συμπεράσματα αυτά για τη βελτίωση της διαχείρισης του χώρου Σέγγεν, διότι νομίζω ότι αυτή η έκθεση εξυπηρετεί άριστα αυτό το σκοπό. Όσον αφορά τα προσωπικά μου συμπεράσματα από την έκθεση, υπάρχει μόνο ένα θα έλεγα. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν ανέφερε σαφώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το εξής. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και λιγότερο σοβαρά προβλήματα όσον αφορά το κεκτημένο Σέγγεν σχετικά με την αστυνομική συνεργασία, σχετικά με το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν και πώς λειτουργεί αυτό και σχετικά με σφάλματα που περιέχουν εκθέσεις των κρατών μελών. Για να διορθωθούν όλα αυτά τα προβλήματα, Δεν είναι απαραίτητο να εργαζόμαστε συγκεκριμένα ρητά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Χρειαζόμαστε ένα νέο μηχανισμό για να ανακαλύπτουμε τα κενά και τα προβλήματα και να βρίσκουμε λύσεις. να μας βοηθήσει να βρίσκουμε λύσεις στο σύστημα. Χθε είδαμε το Συμβούλιο για μία ακόμη φορά που προσπάθησε να υπονομεύσει του νέου συστήματος αξιολόγησης ε, τα κράτη-μέλη στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων προσπαθούν να περιθωριοποιήσουν το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την ε, υιοθέτηση του νέου αυτού μέσου Σέγγεν. Προσπαθήσαμε να το εμποδίσουμε αυτό από το να συμβεί. Τουλάχιστον η Ρουμανία την επόμενη εβδομάδα θα ξανή σημείο της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου και ελπίζω όλοι οι συνάδελφοί μας εδώ να απευθύνουν μια θερμή έκκληση προς όλα τα κράτη-μέλη ούτως ώστε να μπορέσουν να κινηθούν σωστά ε, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. και ελπίζω ότι θα γίνει κάτι για να υποστηριχθεί το δικαίωμα των πολιτών στην ελεύθερη ε, διακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο χώρο Σέγγεν. Διότι αυτό θα πρέπει να γίνει σεβαστό, αυτή είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να τύχει σεβασμού όσον αφορά την άποψή του. Όσον αφορά την ομάδα S&D και την άποψη που έχουμε, όσον αφορά το όλο πακέτο, θέλω να πω ξεκάθαρα ότι εάν το Συμβούλιο παραμείνει αμετακίνητο και θέλει να αλλάξει τη νομική βάση, τότε αποφασίσαμε εμείς να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είμαι σίγουρος ότι όλες οι πολιτικές ομάδες θα μας υποστηρίξουν σε αυτή την προσπάθεια. Για μία ακόμη φορά θέλω να πω ότι αυτού του είδους οι εκθέσεις είναι σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της διαχείρισης του χώρου Σέγγεν και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δουλειά που έκανε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρομέρο Λόπεθ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, είμαστε σε μια δύσκολη στιγμή χρονικά, διότι το Κοινοβούλιο δεν θα δεχθεί ο μηχανισμός αξιολόγησης του Σέγγεν να αποτελεί αποκλειστική απόφαση του Συμβουλίου. Ιδίω όταν είδαμε τελευταία να ομολογεί το ίδιο το Συμβούλιο ότι δεν έχει λειτουργήσει το Σέγγεν. Αν αυτός ο μηχανισμός του Σέγγεν δεν έχει λειτουργήσει και αν αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, είναι δύσκολη αξιολόγηση και είναι δύσκολο να δεχτούμε θα την κάνουν τα κράτη-μέλη. Πρέπει να υπάρχει κοινοτική μέθοδος αξιολόγησης Άρα η κοινοτική μέθοδος εξολόγησης περνάει φυσικά και μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όλες και οι πολιτικές ομάδες θα συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό. Πρέπει να αναλύσουμε την ουσία. Ζούμε σε μια περίοδο που ποτέ το Συμβούλιο δεν είχε τόσους μηχανισμούς ελέγχου. Έχουμε το ΣΥΣ, το ΒΙΣ, αρχεία, πάμπολα για τον έλεγχο των ροών. Και παρόλα αυτά, σε ό,τι αφορά το ανέλεγχο των συνόρων, ε, δεν ε, επιφέρει καμία πρόοδο τόσο συμβούλιο. Είναι σαν ε, να κινείται στα τυφλά. Και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν κάποια συγκυριακά γεγονότα και περιστατικά και δεν μελετώνται, δεν βλέπουμε τι πραγματικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη με τις μεταναστευτικές ροές. Είχα προειδοποιήσει τις προάλλες ότι υπάρχει στη Φλωρεντία Ευρωπαϊκό Ίνδρυμα. Το Τμήμα Μετανάστευσης του Ινστιτούτου αυτού έχει κάνει μια μελέτη για τις 10 ε, μειονότητες, μάλλον πληθυσμούς από τα 27 κράτη-μέλη που μεταναστεύουν. Και στι 10 αυτέ μειονότητε δεν υπάρχει καμία χώρα από την Νότια Αφρική. Άρα αλλού είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ούτε στη Μεσόγειο ούτε στη θάλασσα γενικά. Είναι στι χερσαίε ε, διελεύσεις και στις διαέρος ε, διελεύσεις μεταναστών. Εκεί είναι το πρόβλημα. Από το να έρχονται και από τη στεριά, όχι από τη θάλασσα οι περισσότεροι μετανάστες. Είδαμε επίσης το φαινόμενο της Λαμπεντούζα. Η Γαλλία και η Ιταλία δεν επικεντρώθηκαν σωστά σε αυτό το θέμα. Δεν σεβάστηκαν την νομοθεσία. Υπήρχε η οδηγία προσωρινής προστασίας που δεν δρομολογήθηκε, δεν τέθηκε σε ισχύ ουσιαστικά. Και βέβαια, λόγω της κακής επίλυσης, ε, μετά έγιναν εμβαλωματικές προσπάθειες. Και το μόνο που μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι ότι το Συμβούλιο δεν τα κατάφερε, δεν πέτυχε ούτε στη στρατηγική του να προασπίσει το Σέγγεν, αν πραγματικά αυτός είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή. ούτε να διατηρήσει την ε, στρατηγική αυτή που λέω για την προστασία του Σέγγεν, ούτε και για την αντιμετώπιση των συγκυριακών ε, προβλημάτων που τίθενται και θα συνεχίσουν να τίθενται. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η χρονική συγκυρία. Πρέπει να ακουστεί φωνή του Κοινοβουλίου και να υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη να εστιάσουμε το πρόβλημα εκεί που είναι. Το πρόβλημα δεν έγκυται στην αναστολή του Σέγγεν όταν γίνεται κάτι, όπως αυτό με κεντρική τράπεζα στη Βαρκελόνη μια αθλητική διοργάνωση, όπως στην Πολωνία, Ουκρανία. Ε, τα μεταναστευτικά ρεύματα είναι το πρόβλημα. Και δυστυχώς ε, αυτά τα συγχαίουμε με ροή, ε, με εισρωή μάλλον ε, τον άσυλο. Ε, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το εξεραζόμαστε από αυτή την σκοπιά. Είναι λάθος αυτοί που αναλύουν ή πρέπει να αναλύσουν το φαινόμενο δεν αναλύουν σωστά τα πράγματα. Ας αναλύσουμε πού μπορούν να έγκυνται τα πραγματικά προβλήματα με τις μεταναστευτικές ροές και ο πρώτος ενδιαφερόμενος είναι το Συμβούλιο βέβαια γι' αυτό και μετά η Κομισιόν και μετά το Κοινοβούλιο. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δύο είναι οι ομιλητές Βέμπερ και Σδανόκα τελευταίοι. Κυρία Βέμπερ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την Κομισιόν που ήρθε στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, για να συζητήσει μαζί μας την έκθεσή της αυτή, που πραγματικά είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, θα έλεγα, για τη λειτουργία του Σέγγεν, ε, η διαχείριση του χώρου Σέγγεν αυτούς τους μήνες. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο θέμα και φλέγον, ζέων διότι είναι ένα ζήτημα ε, που ενδιαφέρει την κοινή γνώμη. Όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, ακόμη και, αυτές, και αυτούς που προέρχονται από χώρες που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στη Συμφωνία Σέγγιν. Ελεύθερη κυκλοφορία δηλαδή μέσα στο χώρο Σέγγιν. Γι' αυτό και καλωσορίζω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να μας παρουσιάσει τα πορίσματά της. Το γενικό συμπέρασμα ή μάλλον τα γενικά συμπεράσματα είναι θετικά, αλλά δεν είναι όλα και τόσο τέλεια. Καλό είναι αυτό βέβαια, γιατί δεν μου αρέσει το τέλειο. Το τέλειο με φοβίζει, μπορώ να σας πω. Αν μελετήσουμε αυτά τα δύο παραδείγματα μέσα σε αυτό το εξάμεινο, Είχαμε λόγω της ε, G20 κάποιες ε, διευθετήσεις ε, στην Ιταλία, στην Γαλλία, μετά στη Βαρκελόνη γιατί συνεδρίαζε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πάλι υπήρξαν κάποια μέτρα εκεί στο αεροδρόμιο. Μα υπάρχει κάποιος που φαντάζει ότι κάτι μπορεί να συμβεί επειδή συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και επανισάγει τους ελέγχους στο δρόμο της Βαρκελόνης. Μήπως παρά είναι λίγο αυτό. Μήπως πάει λίγο μακριά. Γιατί πριν από κανένα δύο χρόνια είχαμε ασχοληθεί με πολλά τέτοια θέματα και είχαμε ρωτήσει και την Κομισιόν. Κάθε φορά πια τόσο πολύ δικαιολογείται αυτός ε, η εισαγωγή των ελέγχων. Μήπω στέλνουμε στου πολίτες ένα μήνυμα ότι τους φοβόμαστε. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτός ο νέο μηχανισμό για τον οποίο συζητούμε αυτές τι ημέρε θα πρέπει να συνοδεύεται από μια πιο κοινοτική προσέγγιση και η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα πει το κοινοβούλιο που απαρτίζεται από τους άμεσα εκλεγμένους ερετούς εκπροσώπους των πολιτών. Μήπως θα πρέπει η φωνή του να ακουστεί. Οι συνάδελφοί μου, ο κύριος Κοέλιο και ο κύριος Σέντσο ανέφεραν και μια άλλη πτυχή. Και δει τους μηχανισμούς αξιολόγησης και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επ' αυτού του θέματος όπως προείπαν, είναι απαράδεκτο. Θεωρούμε απαράδεκτο να αλλάξει νομική βάση και όσο μάλλον όταν πιστεύουμε ότι το, Ευρωπαϊκό, το, Συμβούλιο μάλλον δεν έχει παίξει και δίκαιο, σωστό παιχνίδι αν θέλετε. Χθες στις συνεδρίες των συντονιστών ζητήσαμε, και όχι απλά ζητήσαμε, πώς να το πω, Επιφορτήσαμε τον πρόεδρό μας με την υποχρέωση να αποστείλει στο Συμβούλιο μια επιστολή για το τι σημαίνει θεμητή συνεργασία των ε, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θεωρούμε ότι ήταν αθέμητη κίνηση εκ μέρους του Συμβουλίου αυτή. Δεν μπορώ παρά να ελπίζω ότι θα συνειδητοποιήσουν τα κράτη-μέλη ότι έχουν το ίδιο συμφέρον με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι θέλουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Επομένω, η αντιπαράθεση, η ελκυστίδα Κοινοβουλίου-Συμβουλίου για ένα ζήτημα τόσο προσφυλέ προς όλους είναι, πώς να το χαρακτηρίσω, παιδιάστικο, γελίο, σίγουρα πάντως άδικο. Ελπίζω να έρθουν καλύτερε εποχέ και στη... σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του χώρου του Σέγγεν. Ντανόκα, Yes. Σας ευχαριστώ. Συμφωνώ με αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητέ και ιδιαίτερα με αυτά που είπε ο Κάρλος. Είμαι σκιώδης και εγώ για την ε, έκθεση αυτή. Έχει γίνει κάποιος διάλογος με το Συμβούλιο για τις διαφορετικές αυτές ε, προσεγγίσεις. Καλώς ορίζω ιδιαίτερος. Να πω δύο λόγια για τη Λετωνία, το κράτος μου, τη χώρα μου. Ιδιαίτερα επειδή αναφέρεται στη φάση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού. Καλωσορίζω αυτά τα μελλοντικά σχέδια ασφαλώς. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα βρείτε πολύ, πολλά ενδιαφέροντα σημεία. Στα τέσσερα από τα δέκα γεγονότα που αναφέρετε. Αναφέρεται και η Λετωνία. Σας ευχαριστούμε. Στο κεφάλαιο αυτό μιλάτε για την έλλειψη ιστορικών ελέγχων και λέτε ότι έχουν γίνει κάποιες μελέτες και για οκτώ περιπτώσεις Πρόκειται για αστυνομικούς ελέγχους ε, κοντά στα εθνικά σύνορα. My question is when will appear the findings and... Πότε θα βγουν τα απορίσματα, ρωτώ. Μήπως θα πείτε δύο λόγια για το θέμα αυτό. Study. Thank you. Okay, thank you. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Και δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει και η Προεδρία. Um, thanks, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια που κάνετε για την έκθεση. Καταρχάς, ε, επειδή είναι η πρώτη μας έκθεση, καλωσορίζουμε ιδιαίτερως ε, οποιαδήποτε σχόλια, γιατί θέλουμε στο μέλλον να χρησιμοποιήσουμε φυσικά την δομή αυτή, αλλά οτιδήποτε στοιχεία μπορείτε να μας δώσετε είδη σχολείων είναι ευπρόσδεκτα σε ό,τι αφορά και το νομοθετικό πακέτο που αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της βελτίωσης του Σέγγεν. Ο κύριος Κοέλιο ρώτησε κατά πόσο είμαστε απεσιόδοξοι. Κοιτάξτε, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να είμαστε αισιόδοξοι και ρεαλιστές σε σχέση με το τι χρειάζεται για να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση των δραστηριοτήτων που αντιμετωπίσουμε. Και ξέρετε τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η εξέλιξη αυτή και για τον κώδικα για τον και τα σύνορα του Σέγγεν και για το εργαλείο αξιολόγησης του Σέγγεν προκειμένου να καταστούν ε, καλά εργαλεία αποδοτικά στη χρήση τους. Ε, δεν μιλάμε για μία μάχη εξουσιών. Ο διακυβερνητισμό έχει τους περιορισμούς του, αλλά δεν ε, αμφισβητούμε την αρμοδιότητα των κρατών μελών σε περίπτωση που θεωρούν ότι υπάρχει απειλή της δημόσιας τάξης ε, να επανεισάγουν ε, συνοριακούς ελέγχους. Αναμένουμε και σχετική έκθεση από την Ισπανική κυβέρνηση σε σχέση με την επανεισαγωγή τέτοιων μέτρων στη Βαρκελόνη. Πρότασή μας φυσικά δεν θα αλλάξει. Πάντα προτείνουμε τα κρατημέλη να λαμβάνουν την αποφασία αυτή. Γιατί φυσικά ο αντίκτυπος έχει να κάνει και επηρεάζει τους πολίτες όλων των κρατών μελών. Τώρα συγκεκριμένα για τα ερωτήματα που τέθηκαν. Για τις παραβιάσεις. Στη φάση αυτή δεν μπορώ να σας δώσω πάρα πολύ, πολλές λεπτομέρειες. Ίσως ο συνάδελφος να σας πει, ή συνάδελφος να σας πει δύο λόγια παραπάνω για τα θέματα αυτά. Μαριάν Πεζόν με και εγώ επεξεργάζομαι αυτό το θέμα μαζί με άλλους. Να σας πω ότι αυτή η υπόθεση αφορά από τη μια τους αστυνομικούς ελέγχους που ενεργεί η Λετωνία στα εξωτερικά σύνορα και από την άλλη την ομοθεσία της Λετωνίας που αφορά την υποχρέωση να έχει κανείς στην κατοχή του να μπορεί να επιδείξει κάποιο δελτίο ταυτότητα όταν είναι εντό τη επικρατεία και είμαστε σε επαφή με τι αρχέ τη χώρα για να ξεκαθαρίσουμε κάποια ερωτήματα που υπάρχουν και περιμένουμε σύντομα κάποια αποτελέσματα. Σα ευχαριστώ. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Η Προεδρία θέλει να παρέμβει όσον αφορά την νομική βάση και ούτω καθεξής. Απάντηση νομίζω ότι πρέπει εντάχει. Κυ... Κύριος Κοέλιο, κυρία Βίβερ και η ομάδα που εργάστηκε για την Προεδρία συνεργάστηκαν στενά από την αρχή. Γενικός στόχος ήταν να εστιαστούμε επί της ουσίας και μόνο. Το αποτέλεσμα που είναι στο Συμβούλιο τώρα συμπεριλαμβάνει όλες τις θέσεις του Κοινοβουλίου, τις κόκκινες γραμμές μη υποχώρησης, πλήρως ε, ή εν μέρη και είναι καλύτερο το σύστημα αξιολόγηση αυτό που προτείνεται από το ισχύον. Φτάσαμε σαν σταυροδρόμι. Δεν μπορούμε να πετύχουμε ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο για μια νομική βάση σύμφωνα με το άρθρο 77. Είναι ανέφικτο. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε. έχει γίνει μια καινούργια ανάλυση και γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας που όχι μόνο υποστηρίζει τη θέση αυτή αλλά τη διευκρινίζει. Η μόνη λύση είναι είτε να χρησιμοποιήσουμε το 70 ως βάση που ήταν εκεί η βάση είτε να καταπέσει αυτή η πρόταση. Αλλά εφόσον το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν κοινή επιθυμία τη βελτίωση του συστήματος ε, αξιολόγησης δεν βλέπουμε άλλη θεμητή συμπεριφορά από πλευράς Προεδρίας παρά προσπάθεια βελτίωσης του συστήματος. Αυτή είναι η επιλογή, δεν είναι η βέλτιστη για τη συνεργασία μεταξύ των φορέων. Έχουμε καλύτερο προϊόν τώρα όμως από ό,τι κατά το παρελθόν και είναι προ όφελο και των διεθεσμικών οργάνων η εξολόγηση να γίνεται πολύ πιο αποτελεσματικά και πώς να το πω με πιο αληθή τρόπο στο μέλλον και κυρίως για την προστασία του χώρου Σέγγεν. Ευχαριστώ. Ο κ. Κοέλιο θέλει να ξαναμιλήσει. Σύμφωνο σχόλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το άρθρο 70 της συνθήκης προβλεπόταν ως η τελευταία λύση για τους, ε, τα υπόλοιπα θέματα του τρίτου πυλώνα και την, την αξιολόγηση από ομοτήμους. Ε, μετά τα υπόλοιπα ήταν διακυβερνητικής φύσεως. Όπως ανέφερα και στην πρώτη παρέμβασή μου, όταν μιλάμε για το Σέγγεν, δεν μιλάμε για αυτό, μιλάμε για κάτι που κατά την άποψή μας θα έπρεπε να είναι κοινοτική προτεραιότητα, ευρωπαϊκή μέρημνα και κυρίως μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν πρέπει να είναι αντικείμενο διακυβερνητικών αποφάσεων. Θα πρέπει να αναγνωρίσω τις προσπάθειες που κατέβαλε η Δανική Προεδρία, ούτως ώστε να ικανοποιήσει τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε διάφορα σημεία του κειμένου ουσιαστικά η, έκανε προσπάθηση η Ιδανική Προεδρία να πλησιάσει το κείμενο αυτά που θέλαμε εμείς. Το θέμα είναι ποια είναι η αξία, η ουσία αυτής της προσπάθειας αν εφαρμοστεί δυνάμει του άρθρου 70. Ακόμα και αν, που δεν ισχύει αυτό, ακόμα και αν η ιδανική προεδρία τα καταφέρει, πετύχει, να υπάρξει συμφωνία 100% με, τους, με τις διεκδικήσεις του Κοινοβουλίου και εγκριθεί στο Συμβούλιο μπορεί να αλλάξει αύριο, διότι το Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει ούτε στη λήψη απόφαση αποφασίσει ούτε καν δεν μπορεί να συμβουλεύσει, να δώσει συμβουλές αφορά την νομοθετική διαδικασία. αδίποτε ούτως υπήν κέρδη, αδίποτε ούτως υπήν νίκες, διαβεβαιώσεις που μπορούν να μας δοθούν τώρα από το Συμβούλιο, μπορούν να καταστραφούν αύριο την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα, τον επόμενο χρόνο. Γι' αυτό πιστεύω ότι η απόφαση που είναι έτοιμη να λάβω στο Συμβούλιο για την αλλαγή της νομικής βάσεως δεν είναι μόνο ένα βήμα πιστοχώρησης προς τις εποχές της διακυβερνητικές, αλλά είναι και μια κακή απόφαση διότι φωνεύεται η διακυβέρνηση του χώρου Σέγγεν όπως είχε προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως την υπερασπιστήκαμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Προτάσεις γίνονται για να βρεθεί σωστή λύση, να δούμε κατά πόσο είναι χάρη που μας δίνουν τα κάτι μελη η συμμετοχή μας σαν Κοινοβούλιο, είναι δικαίωμα στο σύγχρονο 21ο αιώνα και στη σύγχρονη δημοκρατία του 21ου αιώνα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνω τη συνεδρίαση. Επόμενη συνεδρίαση στις 11 Ιουνίου στο Στρασβούργο, ε, Δευτέρα απόγευμα στις 7. Γεια σας. Καλό απόγευμα.